λέει τον αστυνομικό αυτό μπορεί να είναι η απαρχή μιας θαυμάσιας φιλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάνια και με αυτή την νότα χιούμορ θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έληξε και αύριο 11.30 ώρα θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ τους πάντες και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης το οποίο ε, ε, ε, αναφέρεται σε μία προφορική ερώτηση για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με σπάνιες γέες και δίνω τον λόγο στον κύριο Τσουκαλά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, οι σπάνιες γέες έχουν κέρια σημασία για εκατοντάδες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας αλλά και για την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών. η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις εισαγωγές σπανίων γεών από την κίνα η οποία μονοπολεί το 97% της παγκόσμιας παραγωγής και διαθέτει το 36% των παγκόσμιων οικονομικών αποθεμάτων. η κίνα διαθέτει ισχυρή επιστημονική έρευνα στο πεδίο και έχει επιτύχει αισθητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή κραμάτων και τελικών προϊόντων την ίδια ώρα η βιομηχανία της ευρωπαϊκής ένωσης στερείται τόσο σε πρόσβαση σε πρώτες ύλες όσο και την τεχνογνωσία για την επεξεργασία τους. αν και οι σπάνιες γαίες δεν είναι τόσο σπάνιες όσο μαρτυρά το όνομά τους οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται γύρω στα 10 με 15 χρόνια για την ανασύσταση μιας βιώσιμης γραμμής παραγωγής. η ευρωπαϊκή ένωση αναπτύσσει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τις πρώτες ύλες ωστόσο το πρόβλημα των σπανίων γιών είναι πολύ πιο άμεσο. οι αυξημένες εγχώριες ανάγκες της κίνας και οι προσπάθειές της να περιορίσει τις περιβαντολογικές επιπτώσεις έχουν ήδη ορίσει αυστηρότατους περιορισμούς στις εξαγωγές την ίδια ώρα που η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται. η κίνα έχει θεσπίσει για το πρώτο εξάμεινο του 2011 χαμηλότατα όρια εξαγωγών μειωμένα κατά 35% σε σχέση με πέρσι ενώ ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί αναμένονται στο δεύτερο εξάμεινο. η έλλειψη αναμένεται να εμφανιστεί με ιδιαίτερη ένταση μέσα στους επόμενους έξι μήνες με αυξήσει τιμών των σπανίων γεών αλλά και διατάραξη των γραμμών παραγωγής. οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 2014 θα υπάρχει έλλειμμα 40.000 τόνων σπανίων γεών παγκοσμίω. τα ερωτήματα προς την επιτροπή είναι άμεσα και πιεστικά ποια είναι τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει η επιτροπή μαζί με τους εταίρους της για να εξασφαλίσει οι εναλλακτικές πηγές σπανίων γεών; ποιε είναι οι εξελίξεις της συζητήσης μας με την κίνα και τους διεθνείς μας εταίρους για το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσουκαλά. Δίνω το λόγο στην κυρία Εκ. Αναρωτιέμαι αν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε κάθε πρόκληση είναι ο φόβος της Κίνας και η κατηγορία ότι παρεμβαίνει ε, κρατιστικά. Ε, θα έπρεπε να προωθούμε το ελεύθερο εμπόριο, να προωθούμε την βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την καινοτομία και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες οπλευράς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όχι όμως συσσόρευση, όχι όμως συσσόρευση πρώτων υλών με χρήματα του καταναλωτή. Η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από σπανίζους, ε, σπανίζουσες πρώτες και πόρους. Ε, οι εταιρείε όμως θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διατηρούν αποθέματα ή Όχι τα κράτη. Η αναποτελεσματική χρήση των πόρων θα πρέπει να αποφευθεί. Χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική πρώτων υλών που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές πρόσβασης. Ε, έρευνα, εμπόριο, καινοτομία, κατασκευή υποδομών για την ανάπτυξη των δικών μας πόρων, ε, εφοδιασμός, εξασφάλιση εφοδιασμού και ανακύκλωση. Η Ευρώπη είναι πλούσια σε πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους και στρατηγικά είναι ε, γεωγραφικά κοντά στις, ε, στις χώρες παραγωγής η Ευρώπη έχει την δυνατότητα να, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Χρειαζόμαστε όμως να ενθαρρύνουμε και την καινοτομία και την έρευνα για εναλλακτικέ λύσεις και να βρούμε τρόπους ε, να χρησιμοποιήσουμε ε, άλλες λύσεις έναντι των ακριβών πρώτων υλών που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες να επωφεληθούν από τον εφοδιασμό που μπορούν να παράσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο βιώσιμο. Χρειαζόμαστε δράση στην καινοτομία λοιπόν και στην κατάργηση των εμπορικών φραγμών, όχι συσσόρευση και αποθήκευση πρώτων υλών και χρειαζόμαστε προτάσεις από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γιές. Yes. Και ακόμα δεν έχουν έρθει τέτοιες προτάσεις. Euh, ο τρίτος συντάκτης, ο κύριος Σιμάσκη, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η Υπάρχει το πρόβλημα της ε, ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας αυτής που κινδυνεύουμε να χάσουμε και γι' αυτό δεν πρέπει να παραβλέψουμε κανέναν τομέα, να βασιστούμε στους δικούς μας πόρους, τους οποίους κακώς εγκαταλείψαμε, να στραφούμε προς την εμπορική πολιτική για να μην υπάρχει στρέβλωση του ε, ελευθέρου εμπορίου και να ε, μην ε, βασιστούμε μόνο στην ανακύκλωση η οποία είναι δαπανηρή αυτών των υλών πρέπει να υπάρξουν ορισμένες ερωτήσεις που θα τεθούν σχετικά με την πολιτική των πρώτων υλών. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει την προστατευτική πολιτική της Κίνας επί του θέματος. Δεύτερος, όσον αφορά την ανακύκλωση έχουμε εξετάσει επαρκώς τους πόρους μας τρίτον έχουμε αξιολογήσει την, ε, ε, το κόστος μας και πόσο κοστίζει η ανακύκλωση αυτή ευχαριστώ τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε όπως γνωρίζετε στις αρχές του Φεβρουαρίου η Κομισιόν ανέκρινε την ενημέρωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες. Και αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμφωνίες με την Αφρικανική Ένωση. Έχουμε εντάξει στην ατζέντα των ε, συναντήσεων με την ε, Ρωσική Συνομοσπονδία το θέμα των πρώτων υλών και όπως είπα και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης τον Ιούνιο θα βρίσκομαι στη Βραζιλία στην Αργεντινή και στη Χιλή για να ξεκινήσουμε <laughs> δράσεις διπλωματικές και με αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μετά θα μιλήσω για τις σχέσεις με την Κίνα. Δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση του βιώσιμου αναφοδιασμού μέσα στην Ένωσή μας και γι' αυτό και ενημερώσαμε τις εφαρμοστικές διατάξεις του Natura 2000 σε συμφωνία με τον Επίτροπο Ποτόσνικ γιατί η, έτσι ώστε η ερμηνεία να μην είναι επιζήμια για την εξορρυκτική βιομηχανία ενώ ταυτόχρονα να σέβεται το περιβάλλον. Ο τρίτος πυλώνας αφηρά την ανακύκλωση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και επαναλαμβάνω τα όσα είπα στη διάρκεια της προηγούμενης συζήτηση ότι στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας προβλέπουμε μια σειρά εταιρικών σχέσεων καινοτομία σε διάφορους τομείς. Ο ένας εξ αυτών είναι ο τομέας των πρώτων υλών, όπου η Innovation Partnership βασίζεται στις δραστηριότητες στον τομέα της ε, ανακύκλωσης και της υποκατάστασης των πρώτων υλών. Η νέα ανακοίνωση ωστόσο τονίζει κυρίως η κατάσταση προσφοράς ε, των σπανίων γεών και άλλων βασικών πρώτων υλών. Σύγχρονα, ε, σίγουρα ο περιορισμός των εξαγωγών των σπάνιων γεών περιορίζει φυσικά την παγκόσμια προσφορά. Εξαζιολογούμε την κατάσταση ώστε να εντοπίσουμε τα πιο κατάλληλα μέσα σε πολυμερές επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας εκεί και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις διμερείς μας σχέσεις με την Κίνα στο πλαίσιο του ΠΟΕ έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία επίλυσης διαφορών απέναντι στην Κίνα που αφορά την πρόσβαση στις ε, νέες κύριες πρώτες ύλες το 2009. Εξετάζεται η κατάσταση και η υπόθεση μάλλον και έχει προχωρήσει και η έκβαση θα είναι πολύ σημαντική για το αν θα προχωρήσουμε σε μια άλλη διαδικασία στον ΠΟΕ για τις σπάνιες Τώρα, σε διμερές επίπεδο έχουμε ε, ε, θέσει το θέμα πολλές φορές ε, στην ε, κινέζικη κυβέρνηση σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Το τέλος του 2011 δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας ανάμεσα στην Ένωση και την Κίνα για να διευκολυνθεί ο διάλογος για τα θέματα ε, που αφορούν τις, πρώτες, τις σπάνιες και τις πρώτες ύλες. Έχουμε λοιπόν στρατηγικές ε, εταιρικέ σχέσεις και στις, πρέπει να έχουμε μια δραστήρια διπλωματία για τις πρώτες ύλες με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις ε, πρώτες ύλες, ιδιαίτερα τις πιο σημαντικές. Ένα παράδειγμα, όπως έλεγα, ε, αποτελεί η έναρξη ενός διμερούς διαλόγου στο πλαίσιο της κοινή στρατηγικής Αφρική Ευρωπαϊκή Ένωση 2011-2013 και αφορά μια ειδική, ένα ειδικό τμήμα που είναι αφιερωμένο στις πρώτες και στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Σας τις ανέφερα στο εσωτερικό της Ένωσης εμείς μιλάμε για την ε, ε, ε, έρευνα για τις βασικές πρώτες ύλες. Το πρόγραμμα ProMine είναι αυτό, 2009-2013, στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και όσον αφορά την ανακύκλωση, αυτό αφορά τεχνολογικές προκλήσεις τεράστιες, καθώς η ποσότητα των πρώτων υλών που περιλαμβάνεται σε διάφορα προϊόντα είναι πολύ μικρή. Και η στρατηγική μας έχει στόχο να προωθηθεί η ανακύκλωση μέσω δράσεων που στόχο έχουν την καλύτερη εφαρμογή της ε, νομοθεσίας της ε, Ένωσης για, θέματα, ε, για τα θέματα των αποβλήτων. Επίσης θέλουμε να ευνοήσουμε την έρευνα στον τομέα της ανακύκλωσης και της υποκατάστασης όπως ήδη έχει γίνει στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιου για την χρηματοδότηση προγραμμάτων που στόχο έχουν την υποκατάσταση των σπανίων γεών. Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν αξιολογεί τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια εταιρική σχέση για την καινοτομία στο πλαίσιο των πρώτων υλών και ελπίζει να παρουσιάσει σχετική συγκεκριμένη πρόταση στους επόμενους μήνες. Έχουμε μάλιστα ξεκινήσει και μια συνεργασία με τις ΕΠΑ σε θέματα καινοτομίας και να ερευνούμε τη δυνατότητα συνεργασίας και με την Ιαπωνία. Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στο θέμα των ε, βασικών πρώτων υλών για να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας και να εξασφαλίσουμε ότι ο ανεφοδιασμός μας σε πρώτες ύλες ε, είναι ναι, θέμα των ίδιων των επιχειρήσεων. Όμως θα πρέπει να συζητήσουμε σε στενή συνεργασία με τα κρατημέλη το κόστος, πιθανή, την πιθανή ωφέλεια και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος αποθήκευσης πρώτων υλών. Αυτά κάνουμε. Φυσικά είμαι πάντοτε έτοιμος να ακούσω προτάσεις που προέρχονται από το Κοινοβούλιο, ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε μια δραστήρια δράση της Κομισιόν ε, πάνω στο θέμα αυτό που είναι τόσο σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού ιστού της Ένωσης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρούμπικ από πλευρά του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ταγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία σας γιατί οι πρώτες ύλε είναι η βάση για μια υγιή βιομηχανία του μέλλοντος και γι' αυτό δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την εμπορική πολιτική και να έχουμε διμερείς συμφωνίες όχι μόνο με την Κίνα αλλά και πολλές άλλες χώρες οι οποίες βασίζονται στο να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους αλλά να έχουμε μακροπρόθεσμες συμφωνίες οι οποίες θα αποδώσουν και που θα καλύψουν και τις επενδύσεις για νέα ορυχεία. Όταν υπάρχουν λοιπόν νέα ορυχεία τα οποία ανταγωνίζονται τα ισχύοντα θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν. Σύμφωνα με, την, ε, ε, με τον ΠΟΕ θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε με βάσει στο πακέτο της Σιγκαπούρης το οποίο ήδη έχουμε προωθήσει και θα πρέπει ε, να υπάρξουν παράλληλες διμερείς συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λεπτομέρειες αλλά βλέπουμε ε, σε τι τιμή υπάρχει επεξεργασία κάποια σύλληση στην Κίνα και τι τιμή υπάρχει στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις σπάνιες γεές αλλά και τον μαγνησίτη που είναι ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο, μια πρώτη ύλη ε, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς ε, ούτε να παράγει γυαλί ούτε και πολλά άλλες ε, και πολλά άλλα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα υποκατάστατα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό συμφωνώ με την άποψη του Επιτρόπου Χέλεγκαρτ για το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα το οποίο πρέπει να υπάρχει και βάσει του οποίου να υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που θα επιβληθεί. Ευχαριστώ τώρα κύριε Φρίσκοφς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να ε, υιοθετήσουμε μια μακρόπνοη στρατηγική πρώτων υλών και αποτελεσματική στρατηγική. Οι σπάνιες γεές δεν είναι δεν τη χάνουν μιας εμπορίας όπως άλλα υλικά και άλλες ύλες. Ε, και πολλές φορές οι περιοχές ε, παραγωγής τους, η εξόριξης τους βρίσκονται πολύ κοντά σε ε, πολεμικές ζώνες. Λοιπόν, ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. και βέβαια δεν αρκεί μόνο να παράγουμε τέτοιες ύλες, αλλά πρέπει να τις ανακυκλώνουμε μέσω εφιών διαδικασιών και λογικών στρατηγικών. Είναι εύκολο να εξορίξουμε, αλλά πρέπει να ανακυκλώνουμε κιόλα. Θα πρέπει η ανακύκλωση να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της νοοτροπίας μας. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ρινάλντι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, δώσατε κάποιε υποδείξει, Ωστόσο, θα ήθελα να... κάποιες διευκρινήσει. Καταρχήν, ΠΟΕ, τι κάνουμε ακριβώς στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με την πρωτοβουλία που ήδη αναλάβαμε το 2009 αλλά που από όσο γνωρίζω ε, αφορούσε το μαγνήσιο και το βοξίτη μόνο. Έχουμε μια διαδικασία στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τις σπάνιες γέες. Είναι δυνατόν και το κάνουμε αυτό μόνοι μας ή μπορούμε μαζί με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε όπως θα ήταν ευκταίο. Δεύτερον, είπατε ότι πρέπει να αυξηθεί ο ανεφοδιασμός άλλων και και ευρωπαϊκών. Έχει εκεί ρόλο να παίξει η Γρυλανδία. Τι ακριβώς, ε, ποια ακριβώς είναι η θέση μας. Τρίτη σημείο, ανάκτηση σπάνιων γεών από την ανακύκλωση. Πάμε προς μια ευρωπαϊκή ε, πειθαρχία των, ε, όπως αποκολούνται, ε, αστικών ε, όπως λέγονται. Ε, τέταρτη παρατήρηση για την ανάπτυξη της έρευνας. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις και στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και Ακόμη για το σύστημα αποθήκευσης και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε κοινέ ευρωπαϊκές ε, ε, κανόνες για την αποθήκευση. Τέλος, σε ποιο βαθμό διμερός με την Κίνα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επίπεδου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου και στις διαπραγματεύσεις που τρέχουν για τη νέα ε, συμφωνία συνεργασίας με αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Ρινάλντο και ως Μπουτικόφερ δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σίγουρα βέβαια η εξάρτηση από την Κίνα είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει στρατηγική αδυναμία της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη και κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει, δεν πρέπει να βοηθούμε τους Κινέζους και θα πρέπει να ε, απεξαρτηθούμε από τους ε, Κινέζους. Επίσης δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να ξεκινήσουμε έναν ε, ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεν, αλλά να λάβουμε υπόψη και την Ιαπωνία, διότι η Ιαπωνία επλήγει περισσότερο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πρόσβαση Στι στις σπάνιες ε, σε σχέση με την Ευρώπη και αντέδρασε πολύ αποδοτικά και δραστήρια. Με ένα δισεκατομμύριο χρηματοδότησε ε, την ε, έρευνα για ανακύκλωση και για νέα ορυχεία. Εμείς τι ποσό έχουμε διαθέσει για μια τέτοια εναλλακτική λύση. Το, η βασική σκέψη της πολιτικής μας για τις σπάνιες γεές πρέπει να είναι καινοτομία, αποδοτικότητα των πρώτων υλών και αποτελεσματικότητα διότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα για την ανακύκλωση των σπανίων γεών διότι διαφορετικά ε, δεν το αναφέρουμε καθόλου. Δεν είναι μία λύση που πρέπει να μας απασχολήσει μεθαύριο αλλά αλλά άμεσα διότι οι εταιρείε μας ε, έχουν πρόβλημα η Ρόντια, η Όσραμ και άλλες και ακόμη και η Κίνα αυτή τη στιγμή αρχίζει να επενδύει στα υποκατάστατα των σπανίων γεών γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρχουν ανεξάντλητες πηγές όπως τώρα. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποφεληθούμε και να μην ε, κλαίμε ότι δεν έχουμε ευκαιρίες. Ευχαριστώ κύριε Μπίτι Κόφερ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιόμπορ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι σπάνιες γιές ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικές ε, για την τεχνολογική ανάπτυξη. Άρα σημαντικές και για την ευρωπαϊκή καινοτομία. Η αύξηση της χρήσης τους όμως οδηγεί και σε αύξηση της τιμής τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη 124.000 τόνους, αλλά αυτές οι ανάγκες θα αυξηθούν κατά 50% πολύ σύντομα. Από την άλλη μεριά η Κίνα έχει πρακτικά το μονοπόλιο στο εμπόριο των σπάνιων, γεών. Η Κίνα όμως ανακοίνωσε την μείωση κατά 50% των εξαγωγών της. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις του τομέα βρίσκονται εγκατεστημένες στην Κίνα. Και ε, οι Κινέζοι τις έχουν μπλοκάρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό το μονοπόλιο είναι πραγματικό πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ε, σταματήσει αυτή η πολιτική. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ε, δήλωση στη διάσκεψη της Μαυρίτης να γνωριστεί η χρήση αυτών των στοιχείων για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και κριτήρια βιωσιμότητος. Βέβαια αυτή η συζήτηση γινόταν με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά το ίδιο ισχύει και για την Κίνα και για άλλες χώρες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και πιστεύω ότι χρειάζεται μία διεθνή συνεννόηση κατά τρόπον ώστε η Κίνα και οι άλλοι παραγωγοί να επωφεληθούν από τη μεταφορά γνώσεων για τους ε, μεταλλορίχους για να μπορεί να υπάρξει και επιτόπου επεξεργασία των ε, σπανίων γεών ε, δεν μπορούν απλώς να ε, τις εξάγουν και να μας τις παραδίδουν και θα πρέπει να υπάρχουν ε, τεχνολογίες υποκατάστατες διότι διαφορετικές χρειάζεται πολύ υψηλή επένδυση. Ο κύριος Γκασπάρη για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Σήμερα ε, κάνατε ορισμένες ανακοινώσεις σχετικά με το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους επόμενους μήνες. Το πρόβλημά μου είναι ότι και το 2007 μας είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια ανακοίνωση για τις πρώτες ύλε και τώρα ακούμε και τις ανακοινώσεις των τελευταίων εβδομάδων που μοιάζουν πολύ με τις τότε ανακοινώσεις αλλά πολύ φοβάμαι ότι λίγα συνέβησαν τότε και τώρα ε, θα συμβούν επίσης λίγα διότι πρέπει να επιβάλλουμε την άποψή μας υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους πολύ πιο έντονα εμείς έχουμε απεικιοκρατικές αντιδράσεις ε, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην Κίνα όπου βλέπω πως αντιμετωπίζεται το θέμα των σπανίων γεών και ε, πως εμποδίζει άλλες χώρες να επωφεληθούν οπότε δεν βλέπω τι πρόκειται να συμβεί ε, δεν ξέρω αν φταίει η Γενική Διεύθυνσή σας αν φταίτε εσείς αν φταίει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ποιος φταίει τέλος πάντων ποια είναι τα συγκεκριμένα διαβήματα τα οποία αναλαμβάνονται για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι Κινέζοι είναι πολύ δραστήριοι, περιορίζουν τις εξαγωγές, ε, φορολογούν τις εξαγωγές, μας δημιουργούν προβλήματα. Ξέρετε, ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ποια προϊόντα οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή υπερ τι μέτρα πρόκειται να λεφθούν, πώς θα εμποδίσει να συνεχιστεί αυτός ο ανταγωνισμός. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να έχω μία απάντηση από όλων αυτών. Η κυρία Τικάου για ένα λεπτό. Κύριε Πίτροπε, ε, στοιχεία που χρειάζονται για τα τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τις ε, ε, ανεμογεννήτριες, για τους καταλήτες, οι ε, σπάνιες γέες είναι απαραίτητες για τις ε, νέες μη ρηπαίνουσες τεχνολογίες. Αυτά κυκλοφορούν σε παγκόσμια αγορά, αλλά η αγορά των σπανίων γεών δεν είναι αρκετά διαφανής και ο όγκος των συναλλαγών είναι αρκετά περιορισμένος. Η Ένωση εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την εισαγωγή αυτών των σπανίων γεών, διότι το 90% της παραγωγής γίνεται, ελέγχεται, ελέγχεται από την Κίνα. Ε, μιλάμε για αναδυόμενες οικονομίες, μιλάμε για όλο ένα και μεγαλύτερη διάδοση των νέων τεχνολογιών. Πράγμα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το μέλλον αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση των σπανίων γεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακυκλώσει τις σπάνιες γεές, θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και να βρει υποκατάστατα προϊόντα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ενημερωθεί ο κατάλογος των πρώτων υλών αυτών. Ευχαριστώ. Κύριος Γκέρενς για 1,5 λεπτό. Οι <clears throat> διαπιστώσεις α, της προφορικής ερώτησης αποδεικνύουν <clears throat> μάλλον αποτέλεσμα της σπανιότητας αυτών των Τα κράτη που εισάγουν άλλωστε είναι προφανώ ε, πολύ πιο ευάλωτα από τα κράτη που παράγουν αυτέ τι χιλιές. Οπότε θα πρέπει να δράσουμε με δύο τρόπου. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παραμείνει όμοιρος ε, και θα πρέπει να δράσει στο G20, στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΠΟΕ κλπ. Και δεύτερον, θα πρέπει να δράσουμε στο πλαίσιο τη στρατηγική Λισαβόνα για την μείωση τη εξάρτησή μα από τι σπάνιε γιέ σύνθημά μας θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ανακύκλωση και προώθηση της έρευνας για την παραγωγή ε, προϊόντων υποκατάστατων προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε να λαιλατηθούν ή ε, να λαιλατεί το υπέθαφος των χωρών, των αναπτυσσόμενων χωρών. Κύριε η κατάσταση είναι σαφής. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τον εφοδιασμό με σπάνιες γηές, αλλά ο ανταγωνισμός είναι όλο και πιο έντονος. Η Κίνα ελέγχει το 95% της παγκόσμιας παραγωγής και η συνεχής, ε, μείωση των εξαγωγικών ποσοστώσεων ε, έθεσε το θέμα αυτό, τοποθέτησε το θέμα αυτό στην ατζέντα του G20. Το θέμα λοιπόν είναι αποφασιστική σημασία για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η απάντηση θα είναι η συνεργασία με τις χώρες που διαθέτουν αποθέματα, αλλά και μέσω της ανάπτυξης έρευνας και της καινοτομίας. Θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν σε έρευνα και ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές τεχνικές εξόριξης, χρειάζεται να αναζητήσουμε ε, υποκατάστατα για να μειώσουμε την εξάρτηση και βέβαια να προωθήσουμε την ε, ε, ανακύκλωση. Ε, τη, γι' αυτό το λόγο συγχαίρουμε τον κύριο Τατζάνη για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τα επόμενα βήματα της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο ΚΑΤΣΙΑΙ. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανησυχώ πολύ για ορισμένες ε, πράγματα που έχω ακούσει εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ και κάποιες εβδομάδες. Σήμερα ήταν ε, η έλλειψη των σπανίων γεών, πριν από λίγο οι πρωτενε, μετά κλείσανε τα εργοστάσια της ζάχαρης, έχουμε έλλειψη ζάχαρης. Μα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να προωθήσει την βιομηχανία της πια. Ε, φυσικά και καλωσορίζω την δέσμευση του Επιτρόπου να εξετάσει την καινοτομία όσον αφορά την υποκατάσταση κτλ. Επίσης ανακύκλωση και πάνω απ' όλα νομίζω νέες τεχνολογίες. Εγώ παρακολούθησα ένα σεμινάριο πριν από, δύο, από λίγες εβδομάδες στη Βρυξέλλες για την νέα τεχνολογία ε, που έχει αναπτυχθεί για να βρεθούν ε, στοιχεία από το βυθό της θάλασσας. Είναι καλό να πάει βέβαια ο Επίτροπος στη Βραζιλία να συνομιλήσει με την Κίνα, αλλά αν η διπλωματία αποτύχει και δεν μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε, τι θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε σειρή οικονομία θα είμαστε και πολιτικά δύναμη. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ο κύριος Μπαλσίτης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, το θέμα αυτό τον πρώτων έχει άμεση σχέση με την πρόοδο της Ευρώπης και χαιρετίζω την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος αλλά δεν πρέπει να σκεφτούμε μόνο πόσο θα έχουμε πρόσβαση σε πρώτες ύλες στο μέλλον αλλά πώς θα αναπτύξουμε μια οικονομία στην Ευρώπη η οποία θα αποβλέπει στην πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των πρώτων υλών. Η ανακύκλωση είναι η λέξη κλειδί εδώ και θα πρέπει να υπάρξουν και επαρκείς επενδύσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγωγές αυτών των σπανίων γεών θα μας καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς και θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπης του 2020. Αυτή η συζήτηση ε, συνδέεται με την ε, εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και τη συστημική κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Η κρίση που μας ανακοίνωσαν ως χρηματοοικονομική είναι πολύ πιο πλατιά και πιο παγκόσμια. Ε, έχει σχέση με, το, το, την οικονομική ανάπτυξη του καπιταλισμού και το γεγονός ότι ο πλανήτης η Γη είναι γενόδωρος αλλά έχει τους περιορισμούς του. Ε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια και αυτό αποτελεί και την, ε, την, τον περιορισμό του καπιταλισμού. Η φύση έχει τα όρια της. Η εξέλιξη προς ένα πολυκεντρικό κόσμο ε, από οικονομικής και πολιτικής πλευράς ανοίγει το δρόμο για τον ανταγωνισμό για τις πρώτες ύλες. Δημιουργεί συγκρούσεις ε, και η συναλλαγματική και εμπορική πόλεμη, που βλέπουμε είναι συμπτώματα αυτών των συγκρούσεων. Και ε, έχουμε και άλλους, και άλλους συγκρούσεις για το μέλλον. Και βασικά μιλάμε και για αυτά όταν μιλάμε για το θέμα των σπανίων γεών. Ευχαριστώ. Χέρτζοκ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Τώρα τα λέω στα αγγλικά. Όταν γεννήθηκε η γιαγιά μου, ήταν μία από τα δύο δύσει που ζούσαν στη γη. Εγώ όταν γεννήθηκα ήμουν μία από τα πέντε δύσει που κατοίκων τη γη. Και όταν θα γεννηθεί η δική μου εγγονή θα είναι μία από τα εννέα δύσει που θα ζουν στην γη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν νέε τεχνολογίες. Ε, θα ήθελα να... Θυμίσω κάποιον που πριν από 100 χρόνια πήρε το βραβείο Νομπέλ για τη χημεία για τον διαχωρισμό και την ε, καθάριση του ραδίου και του πολωνίου, την κυρία Σκραμπόφσκα, γνωστή ως ε, Μαρία Κιουρί. Χρειαζόμαστε πολλές ε, Κιουρί, πολλούς επιστήμονες, νέες τεχνολογίες και γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω εσάς κύριε Πίτροπε να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε η χημεία να, να χρησιμοποιήσετε τη χημία για να δημιουργήσετε χώρο για νέα ταλέντα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να εισάγουμε τις πρώτες ύλε, αλλά θα μπορούσαμε να τις διατηρήσουμε εδώ ή να τις κατασκευάσουμε βεβαίως με νέες συνεργασίες και με υποκατάσταση. Και πολύ σωστά είπαν συνάδελφοι ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις πρώτες ύλε στην Ευρώπη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συγκέντρωση πρώτων υλών και να δημιουργήσουμε πρότυπα σύμφωνα με τα οποία ε, θα υπάρξει μεγαλύτερη ανακύκλωση και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι το εξής. Θα πρέπει αυτές οι σπάνιες γεές να χρησιμοποιούνται όπου είναι πιο χρήσιμες διότι όσο πιο ε, σπάνια καθίστανται τα μεταλλεύματα ε, τόσο πιο ξύνε το ερώτημα που τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή ε, δεν αξίζει να, υπάρχει, να χρησιμοποιηθεί σε ένα παιχνίδι του McDonald's αλλά ε, σε μια ηλεκτροπαραγωγική μονάδα. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γκίρεκ οι επενδυτές ε, ζητούν ε, γρήγορη, γρήγορα κέρδη και αυτό ε, επηρεάζει και τους καταναλωτές. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μεγάλους επενδυτές που πολύ συχνά έχουν και το μονοπόλιο και αυτοί ορίζουν και τους, ε, καθίζουν και τους όρους. Οπότε η Ευρώπη ε, δυσκολεύεται να αναπτυχθεί εξαιτία ε, έλλειψη σπανίων γεών που είναι απαραίτητε για την παραγωγή, για παράδειγμα στην παραγωγή ολικής ενέργειας κλπ. Οπότε Ήρθε η ώρα να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια του, του εφοδιασμού, του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μιλάμε μόνο δηλαδή για τις σπάνιες γης. Έχουμε και άλλου είδους ε, ορυκτά τα οποία είναι σημαντικά για τους καταλύτες, το βολφράμιο, το λίθιο, το σελήνιο και άλλου είδους ορυκτά. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Γκυρέκ. Με συγχωρείτε, είμαι και εγώ λίγο κουρασμένη. Κύριε Πίτροπο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ο ίδιος... Ναι, δεν είμαι και σε μεγάλη φόρμα. Όλοι κουρασμένοι είμαστε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί με αυτή τη συζήτηση δίνει ισχύ στη δράση που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η δεύτερη Επιτροπή Βαρόζο έχει ξεκινήσει για να λύσει αυτό το λεπτό ζήτημα των σπανίων πρώτων υλών. Όπως σωστά υπογράμμισε ο κ. Σόλτ, από την συνάντηση της Μαδρίτης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια αποφασιστική δράση, όχι μόνο λόγια δηλαδή, αλλά συγκεκριμένε ενέργειες. Και όταν μιλώ για συγκεκριμένες ενέργειες, μιλώ για την επεξεργασία ενός καταλόγου 14 πρώτων υλών σπανίων, και επί των οποίων πρέπει να δράσουμε έναν κατάλογο που φοβούμε ότι δυστυχώς θα χρειαστεί να γίνει λίγο μακρύτερος ε, πρώτο συμφωνία, η πρώτη συμφωνία με την Αφρικανική Ένωση μετά από πολλούς μήνες δουλειάς και που οδήγησε σε μια συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας βλέπουμε την Αφρική να ενδιαφέρεται άμεσα σε κοινή, για κοινή δράση με τη δική μας Ένωση με την Επιτροπή τόσο για τα όσο μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Ένωση, για ανάλυση δηλαδή των αναγκών μας, όσο και για μια ανάλυση των ε, πραγματικών δυνατοτήτων ε, για εξορρυκτικές δραστηριότητες στην Αφρική, την ενδεχόμενη δημιουργία μιας γεωλογικής υπηρεσίας και το πρόγραμμα για τη δημιουργία διαφρικανικών δικτύων εκεί όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί η εξορρυκτική βιομηχανία στην Αφρική. Εκεί. Επίσης ε, με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία δεύτερη φορά συζητάμε για συμφωνίες σε θέματα πρώτων υλών και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο με ανακοίνωση, δυο ε, συναντήσεις έχουν γίνει. Και όπου το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρώτες ύλες δεν είναι ανακοίνωση, αλλά είναι ένα κείμενο εγκεκριμένο από την Κομισιόν, όπου υποδεικνύεται μια σαφής και συγκεκριμένη στρατηγική, όπως σας είπα, που βασίζεται σε τρεις συγκεκριμένους πυλώνες, επί των οποίων σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Η απόφαση για ένα Innovation Partnership ε, που συνδέεται με δράση που θα συμμετέχουν οι ιδιώτες και εύχομαι και το Κοινοβούλιο και οι άλλοι, τα άλλα θεσμικά όργανα για την κοινοτομία και την έρευνα για τον εντοπισμό ισχυρών στεναρών δράσεων για την ανακύκλωση και την υποκατάσταση και αυτό δεν είναι μόνο ανακοίνωση, είναι συγκεκριμένη ενέργεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα αίτημα το οποίο εγκρίθηκε από το σύνολο των Επιτρόπων και άρα αποτελεί τμήμα τη Στρατηγική Επιτροπή όσον αφορά την ε, καινοτομία. Όσον αφορά το θέμα του ΠΟΕ, φυσικά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να λύσουμε με διπλωματικές ενέργειες το θέμα. Η μετάβαση στην Λατινική Αμερική είναι άλλη συγκεκριμένη δράση. Δεν είναι απλώς ανακοινωθέν γιατί τα, οι, οι σε τέτοια λεπτά ζητήματα απαιτούν ε, και πολύ προσεκτική προετοιμασία για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Φυσικά θα παραλείψω να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για τα όσα επιτύχαμε. Όσον αφορά τώρα την πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούμε να δούμε αν οι πρώτες που βρίσκονται στο υπέδαφος, όπως στη Γρελανδία ή στα στενά Μπάρεντς ή σε άλλα μέρη της Βόρειας Ευρώπης θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν η εξορυκτική δραστηριότητα είναι δυνατή, αν είναι σκόπιμη Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν ε, ε, δεχόμενες ερευνητικές δράσεις. Την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, θα γίνει μια πολιτική και τεχνική συζήτηση για τις ε, ευκαιρίες που υπάρχουν στη θάλασσα Μπάρεντς όπου θα συμμετέχουν διάφοροι Σουηδοί υπουργοί μαζί με εμπειρογνώμονες για να αξιολογήσουν αν οικονομικά συμφέρει ή όχι. Και περιβαλλοντικά συμφέρει, γιατί γι' αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Αν πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα εκεί κοιτάσματα. Τώρα για το βιομηχανικό και εμπορικό τομέα ο Επίτροπος Δεγκούχτ είπε επίση ξεκάθαρα πως σκοπεύει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα το κείμενο τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωση στην παράγραφο 5 σημείο 2 το λέω γιατί μπορεί αυτό να ενδιαφέρει και τον ε, κύριο Κάσπαρη που νομίζω έθεσε το ερώτημα αυτό στην ανακοίνωση για τι πρώτε ύλε, παράγραφο. 5.2 γίνεται λόγος για, δυνατές, ε, για, για τις δράσεις αντι-dumping και για δράσεις ε, από εμπορικές, από εμπορικές δράσεις. Ναι, να επαναλάβω σε παράγραφος 5 σημείο 2 για την ανακοίνωση για τις πρώτες ύλες. Αν θέλετε να σας το δώσω. Θα το έχετε ξανά αύριο το πρωί. Όσον αφορά τώρα τις ενέργειες στον ΠΟΕ, για τις οποίες είναι υπεύθυνο ο Επίτροπος Ντεγκούχτ, όπως σας είπα και στην παρέμβασή μου, ξεκίνησε μια διαδικασία με το Μεξικό και τις είπα για τις νέες ε, πρώτες ύλε για να, που περιλαμβάνουν και τις προ, ε, σπάνιες Έχει προχωρήσει το θέμα, κοντεύει στην επίλυσή του και τα απορίσματα θα είναι καθοριστική σημασία για να καταλάβουμε και εμείς στην Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίε θα πρέπει να αναλάβουμε για το θέμα των σπανίων γεών. Αξιολογούμε την κατάσταση ακριβώς για να δούμε ποια είναι τα πιο κατάλληλα μέσα στον τομέα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ανακύκλωση των Ισπανίων γεών και το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ρινάλντι στη διάρκεια της παρέμβασής του, μπορώ να σας πω ότι για την δράση της ανακύκλωσης, αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θα έλεγα ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καλύπτεται το 40% των αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση και η Κομισιόν πρότεινε την σημαντική αύξηση της ε, πρόταση δηλαδή του Επιτρόπου Ποτόσνικ, όχι δική μου, να αυξηθεί η ανακύκλωση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων που, περιέχουν οι σπάνιες γεές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η δράση για τα προϊόντα και με στόχο να διευκολυνθεί η ανακύκλωση στο τέλος της ζωής αυτών των συσκευών. Ήδη υπάρχει μια σχετική νομοθεσία που προετοιμάζεται και ο Επίτροπος και σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και όσον με αφορά, όσον αφορά δηλαδή τη δράση της βιομηχανικής πολιτικής σε σχέση με τις πάνιες γέες και τις πρώτες ύλες, σκοπός μου είναι να προχωρήσω, να μην κάνω υποσχέσεις γιατί δεν είμαι συνηθισμένος στις υποσχέσεις, είμαι συνηθισμένος στο να τηρώ τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνω, κυρίως αυτές που αναλαμβάνω ενώπιον του Κοινοβουλίου, όπως έχω πράξει από τη στιγμή όπου ανέλαβα και μάλλον ε, είχα την εμπιστοσύνη των επιτροπών ενώπιον των οποίων ε, παρουσιάστηκα. Σκοπεύω λοιπόν να προχωρήσω και να τηρήσω τις δεσμεύσεις που ανέλαβα χωρίς να κάνω ανακοινώσεις αλλά προσπαθώντας να δώσω συγκεκριμένε απαντήσεις στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών και σε αυτόν τον λεπτό τομέα της, ε, του ανεφοδιασμού του βιομηχανικού τομέα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα καλά νέα, για τις δεσμεύσεις που θα παρακολουθούμε πέρα τη συζήτηση. Και καλό τον Επίτροπο Έτιγκερ να έρθει κοντά μας και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το καλύτερο το κρατούσαμε για το τέλος, έχουμε τη δήλωση της